30 ψήφου διαφορά. Στην οθόνη μου ήταν απόλυτα σαφέ. Λυπάμαι που δεν έγινε αυτό. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες να το ελέγξουν ώστε στην επόμενη ψηφοφορία να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και όλοι οι βουλευτές να μπορούν να διαβάσουν το αποτέλεσμα στην οθόνη. Θα μπορούσαν οι υπηρεσίες να κάνει το απαραίτητα. Ευχαριστούμε κυρία Μπέρες. Λοιπόν, είπαμε, πρέπει να ψηφίσουμε την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτρόπων βάσει τη πρόταση που παρουσιαστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων. Παράγραφο 1 σημείο 3 αφορά την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Εκεί έχουμε την τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. Ποιο απέ, απέχει. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η απόφαση στο σύνολό τη. Ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε. Η ημερησία διάταξη ορίζεται όπως αποφασίστηκε. Ora, giorno. Τώρα η ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ένα διαδικαστικό. Εγώ δεν βλέπω να λειτουργεί εδώ το μηχάνημα για, το, για την ομάδα του UKIP, το φωτάκι. Θα παρακαλούσα να ζητήσω από τις υπηρεσίες να το τσεκάρουν. Συγγνώμη, το καμπανάκι δεν λειτουργεί στα γραφεία του UKIP. Βεβαίω. Θα στείλουμε κάποιον αρμόδιο για να ελέγξει για να ελέγξει τα τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένω υπάρχουν. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τι δηλώσει Συμβουλίου και Επιτροπή για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τη Μαλτέζικη Προεδρία. Ευχαριστώ.